El Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να καταλάβετε τη θέση σας γιατί αρχίζουν ψηφοφορίες. Ορίστε, κυρία Χάση, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σχετικά με τη σημερινή σειρά των ψηφοφοριών, έχουμε λάβει ένα κατάλογο και το ψήφισμα για τα ε, κριτήρια για την ανάκτηση χάρτου είναι άρθρο 88 η διαδικασία που σημαίνει ότι απαιτείται ειδική πλειοψηφία για να αποφασίσει το Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό φρονώ ότι δεν είναι σωστό που το έχετε βάλει τελευταίο θέμα στις ψηφοφορίες. Κανονικά θα πρέπει να μπει μετά τις υπόλοιπες νομοθετικές ψηφοφορίες που σημαίνει μετά την έκθεση γκρότε ε, για το backloading. Εκεί θα πρέπει να μπει αυτή η τελευταία έκθεση. Και προτείνω το ψήφισμα αυτό λοιπόν να ψηφιστεί μετά την έκθεση γκρότε. Είναι για το ανακτημένο χαρτί που πάβει να αποτελεί απόβλητο. Μάλιστα, κυρία Χάση. Διαφωνεί κανείς με την πρόταση της κυρίας Χάση. Αν όχι, θα ψηφίσουμε όπως προτείνει η κυρία Χάση. Λοιπόν, έκθεση Berlinguer και Κλάις. Πρόγραμμα δικαιοσύνη για την περίοδο 2014-2020. Ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Γκιόνς. Πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια, περίοδος 2014-2020, άρχεται ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Βίνκλερ. Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση Βίνκλερ. Έκθεση Φράγα. Πρωτόκολλο Συμφωνία Αλληλευτική Σύμπραξη Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκου. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. La recomendación. Σύσταση Steinruck. Σύμβαση της ΔΟΕ για την ασφάλεια κατά τη χρησιμοποίηση χημικών προϊόντων στην εργασία. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Σύσταση Ματιέ Ουγιόν. Καταπολέμηση τη παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων. Ψηφί υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ, φωνές από κάτω. Ας το ελέγξουμε λοιπόν. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Σύσταση Σόλτς για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Σύσταση Μορέιρα. Εισαγωγή βοιου κρέατος. Ψηφίπε. Κατά. Επαναλαμβάνει η ψηφοφορία. Δεν σηκώνεται χέρια. Λοιπόν, σύσταση Μορέιρα, επαναλαμβάνω, για τις εισαγωγές βοηού κρέατος. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σύσταση Κοτινή. Πρωτόκολλο Συμφωνίας Αλληλευτικής Σύμβραξης με την ακτή Ελεφαντοστού. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση ΜΑΤΟ. Εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλίας της Καναρίους νήσους. Ονομαστική είναι η ψηφοφορία και αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση να ράχω. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Νέισκι. Το ίδιο θέμα για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Άρχη της ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Κοσλόφσκι. Το ίδιο θέμα πάντα. τη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκθεση Γέγλε. Διαπραγματεύσεις για μια στρατηγική συμφωνία με τον Καναδά. η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Swimborn Πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίασης για τα μη πιστωτικά ιδρύματα. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκθεση νίβλε. Η διαστημική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκθεση Δελκαστήγιο. Υπολογιστικό νέφος ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκθεση σε εδώ. Έκθεση εξολόγησης του Μπερέκ. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκθεση Ρόντουστ. Κοινή ελευτική πολιτική. Η τροπολογία παριθμών 1. Τμήμα πρώτον γιατί είναι κατά τμήματα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου, με προκειμένο. Έκθεση Στίβενσον. Κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Χωρίς τροπολογία. Εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου, λοιπόν. Έκθεση Αρσένη. Βορειοατολικός Ατλαντικός από θέματα βαθαίων υδάτων και αλία σε διεθνή ύδατα. Λοιπόν, 131 τροπολογίες έχουμε της αρμόδιας επιτροπής. Θα τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 29 ε, τροπολογία κατά τμήματα. Τμήμα πρώτον ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 62, ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες. Και τώρα θα ψηφίσουμε την 131. Ψήφιπε... κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία πέρας δεν κρίνεται και καταπίπτει η επόμενη ψηφίζουμε τώρα την πρόταση της Επιτροπής Υπέ. κατά αποχές εγκρίνεται. Και το σχέδιο... Ορίστε. Ο κύριος Αρσένης έχει το λόγο, παρακαλώ, κύριε Αρσένη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βάσει το άρθρο 57 εδάφιο 2 του κανονισμού θα ήθελα η τελική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα να αναβληθεί και να δοθεί η εντολή στην Επιτροπή μας να αρχίσει διαπραγματεύσεις για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτό που πρότεινε ο κύριος Αρσένης. Ψηφίπε. Α, ορίστε κυρία Φράγα παρακαλώ. Πείτε μου. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος πολιτικής μου ομάδας ζητώ να ψηφιστεί τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Το Κοινοβούλιο, οι περισσότερες πολιτικές ομάδες έχουν υπογράψει ένα συμβιβασμό που βλέπετε ότι υποστηρίζεται από την πλειοψηφία. Δεν υπάρχει λόγος αναβολής τελικής ψηφοφορίας. Εχθές μποϊκόταρε το συμβιβασμό εισηγητή, σήμερα έχασε στην Επιτροπή Αλίας είχε την υποστήριξη της πλειοψηφίας ο συμβασμός και προτείνω να προχωρήσουμε στην ψήφιση του νομοθετικού ψηφίσματος. Ο Πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει κυρία Φράγα, σύμφωνα με τον κανονισμό, αυτό που μας πρότεινε ο κύριος Αρσένης πρέπει να ψηφιστεί. Αν θέλετε, αν θέλει το σώμα να ακολουθήσει εσά θα καταψηφίσει. Αλλά πρέπει να θέσω σε ψηφοφορία αυτό που ζήτησε ο κύριο Αρσένης, έτσι κι αλλιώ. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση του εισηγητού, του κυρίου Αρσένη, υπό την εξή έννοια. Ζητεί αναβολή της τελικής ψηφοφορίας. Ψήφι υπέρ τη προτάσεω του κυρίου Αρσένη. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται την πρόταση του κυρίου Αρσένη. Τσεκ φωνές από κάτω. Εντάξει, εντάξει, θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. I think Πέρας. Απερίφθη η πρόταση του κυρίου Αρσένη. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε συνεπώς το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Σε Εγκρίνεται η πρόταση. Περνάμε τώρα στην έκθεση Γκαρντίνη για το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ψηφίζουμε το μπλοκ 1 των τροπολογιών υπέρ παρακαλών κατά, αποχές εγκρίνονται. Ε, καταπίπτει το δεύτερο μπλοκ, ψηφίζουμε το σχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί. Διακόπτει ο πρόεδρος. Ναι, την πρόταση επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προτείνουμε την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που έχει δύο τροπολογίες, 107 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε την τροπολογία 108 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική κλίση, η οποία και αρχίζει. Σε Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψήφια. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Σάντσες Πρεζέδο. Συμβάσεις πίστος για ακίνητα κατοικίας. Τροπολογία 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Και την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική κλίση, η οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Murphy για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές. Το πρώτο μπλοκ τροπολογιών 1 έως 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Και ψηφίζουμε την τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 13 αρχίζει η ψηφοφορία. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπάρχουν 13. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση Επιτροπής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το ψήφισμα, το νομοθετικό ψήφισμα. Ναι, έχετε το λόγο. Ο κύριος Μέρφυ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε με βάση το άρθρο 57 παράγραφος 2 θα ήθελα να μην ψηφίσουμε για, τον, για την νομοθετική έκθεση, ψήφισμα μάλλον, και να γίνει αναπομπή στην Επιτροπή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ο πρώτος τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να γίνει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Θα ψηφίσουμε την πρόταση του κυρίου Μέρφη. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Άρα, περνάμε στην επόμενη έκθεση, που είναι η έκθεση Γκρότε για τον χρόνο διεξαγωγής πληστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής. Ψηφίζουμε απευθείας την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα, σύμφωνα με το αίτημα της κυρίας Χάση, θα ψηφίσουμε την πρόταση ψηφίσματος για την ανάκτηση του χαρτιού. Σύμφωνοι. Ψηφίζουμε καταρχήν την ε, τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος για τα κριτήρια για να ορίσουμε πότε το ανακτηθέν χαρτί ε, δεν ε, αποτελεί απόρριμα. Κυρία Μαγκίνες. Η κυρία Μαγκίνες ζήτησε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας βοηθήσω γιατί πρόκειται για την τελευταία σελίδα του κατάλογου ψηφοφοριών. Δεν ξέρω αν είναι απόλυτα σαφές. Είναι τελευταία σελίδα. Ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια, ε, κυρία Μαγκίνες, στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Ξέρετε τι ψηφίζουμε. Ωραία, θαυμάσια. Γνωρίζετε όλοι τι ψηφίζουμε. Τροπολογία υπαριθμών 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ε, ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Με πολύ μικρή διαφορά απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, ωραία. Ας ελέγξουμε την 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέντε. Ψηφίζουμε την πέντε υπέρ κατά, αποχές. Ωραία, σε ελέγξουμε και πάλι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. Οκτώ. Αρχίζει η ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος, αλλά διορθώνει. Ψηφίζουμε. 8. Υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. 7. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 7. Πέρας. Απορρίπτεται. Οκτώ. Οκτώ τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε και πάλι αρχίζει η ψηφοφορία για την οκτώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε και πάλι. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 9. Πέρας. Εγκρίνεται αυτή τη φορά. Και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της. Περνάμε στην ονομαστική κλίση απευθείας, η οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία, θα διακόψουμε τώρα. Ε, ο κύριος Αλαφράνκα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να διακόψω, ήθελα απλώς να πω ότι δεν ε, ε, λειτουργήσε το μηχάνημά μου όταν ψηφίσαμε την έκθεση Φράγα και υπερψήφισα. Ωραία, αποκαταστάθηκαν τα πράγματα. Τώρα θα διακόψουμε την ψηφοφορία για την ε, πανηγυρική συνεδρίαση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Μαλή και στις 12.30 θα συνεχίσουμε με την ψηφοφορία.